Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, στην Επιτροπή μου είπε ένας, ε, ο, ένας ομιλητής ότι έχει πολύ λίγους φίλους το ISDS στην Ευρωπαϊκή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι αμφιλεγόμενο το ISDS η διαδικασία διαμεσολάβηση μεταξύ επενδυτών και κρατών για πολλούς λόγους. Έχει πολλές συνέπειες για τις δημόσιες υπηρεσίες και τους δημόσιους προϋπολογισμούς. Είναι και μια επίθεση στην δημοκρατική ελευθερία. Αλλά αυτή τη στιγμή το κύριο πρόβλημα είναι η έλλειψη διαφάνειας. Οι διαδικασίες είναι πάντα και κλεισμένων των θυρών και απόλυτα αδιαφανής. Γι' αυτό δεν είναι παράξενο ότι αυξάνεται ο σκεπτικισμός έναντι του ISDS. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ζητήσει στα πλαίσια μια συζήτηση για το TTIP να υπάρξουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε σχέση με το ISDS. Η κίνηση για νέες συμφωνίες περιλαμβάνει αυτό το πρόβλημα, αλλά αυτό ισχύει, το ίδιο πρόβλημα ισχύει για πολλές από τις παλιές συμφωνίες που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου υπάρχουν ρήτρε για τη διαμεσολάβηση αυτή, το ISDS, που είναι απόλυτα αδιαφανή στη διατύπωσή τους. Και υπάρχουν και εσωτερικές αντιφάσεις. Από τη μία πλευρά το Συμβούλιο τονίζει ότι είναι απαραίτητο να έχουμε διαφάνεια σε όλους τους δυνατούς χώρους, αλλά όχι στις συνθήκες τελικά από ό,τι φαίνεται. Σε ό,τι αφορά διμερείς συμφωνίες ISDS είναι όλα κλειστά και επτασφράγιστα. Αυτό είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Ε, γιατί εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή πρωταθλητές της σύναψης συμφωνιών για διαμεσολάβηση μεταξύ επενδυτών και κρατών. Υπάρχει η σύμβαση του Μαουρίτσιους που έχει <clears throat> υποστηριχθεί από τα Ηνωμένα Έθνη και η οποία απαιτεί να υπάρξουν κάποιες προδιαγραφές για τις ε, διαμεσολαβητικές αυτές συμφωνίες. Και αυτό το οποίο τονίζει ο ΙΕ είναι η ανάγκη διαφάνειας για τη χάρτα ενέργειας και που είναι η μόνη περίπτωση όπου προβλέπεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετέχει ως Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από τις συνήθειες της Σαββόνας. Και η υποστήριξη των κρατών μελών είναι ένα δείγμα υποστήριξης για τη διαφάνεια των διμερών συμφωνιών ISDS. Υπάρχει αυτή τη στιγμή και μία ε, διαμάχη για τις αρμοδιότητες για το ποιος είναι αρμόδιος για τα θέματα αυτά. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, μένω εμβρόντιτος κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, ότι υπάρχει μπλοκάρισμα της υπογραφής αυτής της ε, συνθήκης των Ηνωμένων, Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών και από, τις, και από την Κομισιόν και από τα κράτη-μέλη και αυτό δίνει το μήνυμα στον έξω κόσμο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνει πεντάρα για την διαφάνεια και δεν είναι ένας από τους πραγματικούς τους στόχους και πάλι για τη χάρτα ενέργειας κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου. Πολλές φορές αναφέρεται το θέμα αυτό αλλά είναι η περίπτωση που έχουμε τις περισσότερες περιπτώσεις διαμεσολάβησης. 89 περιπτώσεις ISDS. Και αυτό το λέει η γραμματεία του ΟΗΕ για την χάρτα της ενέργειας. Και αυτή τη στιγμή όλα αυτά είναι εν κρυπτό και παραβίστο. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση να δημοσιευθούν τα αποτελέσματα αυτών των ε, ε, διαδικασιών. Τουλάχιστον λοιπόν 89 και μπορεί να είναι και περισσότερες. Αυτή η κατάσταση για μένα είναι απόλυτα απαράδεκτη. Υπάρχουν κάποια, κάτι μέλη που έχουν προσυπογράψει, Γερμανία, Ενωμένο Βασίλειο, Γαλλία, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι. Και γι' αυτό έχω τα τρία αυτά ερωτήματα κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο πιστεύει ότι πρέπει να πείσει τα κράτη-μέλη να ξεπεράσουν αυτή την στάση εμπλοκής και να υπάρξει υπογραφή για την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύει επίσης το Συμβούλιο ότι με τη στάση αυτή εμπλοκής θίγεται και καταρακώνεται η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του εξωκόσμου. <clears throat> Γιατί μιλάμε πάντα για διαφάνεια, αλλά κάνουμε ακριβώς το αντίθετο σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες διαμεσολάβησης. Και το τρίτο ερώτημα μου είναι, θα δώσει κίνητρα το Συμβούλιο, οι Προεδροί του Συμβουλίου να υπογράψουν και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη που δεν έχουν δεχτεί να το κάνουν αυτό, ώστε να είναι σαφέ μέχρι το τέλο του κόσμου, του, του έτου, ότι όλοι υποστηρίζουμε τη διαφάνεια και στι διαδικασίε αυτέ διαμεσολάβηση ε, διαφωνιών. Ευχαριστώ κύριε Λάγκε. Ακολουθεί ο υπουργό Κούντερς τώρα. Uh, ευχαριστώ κύριε Λάγκη. Σας ευχαριστώ για τις τρεις ερωτήσεις σας. Θα μπορούσα να απαντήσω πολύ σύντομα ναι, ναι, ναι. Και θα είχαμε τελειώσει. Αλλά καλό είναι να το έτσι εμπλουτίσω λιγάκι αυτό το αυτή την απάντηση. Τρεις φορές ναι βέβαια. Η διαφάνεια είναι κλειδί για την Προεδρία μας. Είναι μία από τις προτεραιότητες ε, το να εστιάζουμε στα ουσιαστικά απλή και πιο αξιόπιστη νομοθεσία, όπως είπατε. Το Συμβούλιο στα συμπράσματά της για την επενδυτική πολιτική του Νοεμβρίου του 2015 αναγνώρισε ότι σε μια υπεύθυνη εμπορική πολιτική ε, πρέπει να έχουμε υψηλό βαθμό διαφάνεια, πραγματική επικοινωνία με του πολίτε και καλύτερη εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων στην προετοιμασία των διαπραγματεύσεων και εφαρμογή πρωτοβουλειών ε, στον τομέα με σεβασμό των θεσμικών ισορροπιών και των εφαρμοστέων κανόνων. Επομένως, ε, έχετε το δεύτερο ναι. Στα πλαίσια των διαφορών και της επίλυσης διαφορών ε, επενδυτών κρατών, έχουμε κάνει τεράστιε προσπάθειες ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση για να βελτιώσουμε συνολικά το επίπεδο διαφάνειας, όπου υπάρχουν διενέξεις με μέγιστη πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα, σε ακροματικές διαδικασίες και δυνατότητα τρίτων μερών να υποβάλουν έγγραφα. Η Κομισιόν ανακοίνωσε την πρόθεσή τη. να να συμβάλλει με τον κοινοτικό προϋπολογισμό για την αύξηση της διαφάνειας, χρηματοδοτώντας ε, την ε, UNCITRAL και ένα δημόσια προσπελάσιμο μητρό για έγγραφα και προφανώς ε, υποστηρίζει τους κανόνες διαφάνειας UNCITRAL και ISDS. Θέλουμε συστηματικά να ενσωματώσουμε τα πρότυπα διαφάνειας σε όλους τους κανόνες, σε όλες τις ε, συμφωνίες εμπορικές και επενδυτικές που διαπραγματευόμαστε για να διευκολύνουμε την εφαρμογή στις ε, ισχύουσες ε, συμφωνίες ή πολυμερείς συμφωνίες, το είπατε και εσείς που διαπραγματευτήκαμε υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, την σύμβαση του Μαυρίκιου, το Φεβρουάριο του 2014 το Συμβούλιο ε, έδωσε το πράσινο φως στην Κομισιόν για να συμμετέχει σε διαπραγματεύσει αυτής της σύμβασης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σύμβαση θα αφορούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση για μία συνθήκη, δηλαδή την ε, ενεργειακή χάρτα την οποία αναφέρατε. Η απόφαση της Ένωσης να προσυπογράψει την ε, σύμβαση Όπω αναφέρατε και εσεί, αποδείχθηκε δύσκολη. Παρά τι συζητήσει που κάναμε στο Συμβούλιο πέρυσι με βάση των προτάσεων τη Κομισιόν για να ληφθούν αποφάσει για την υπογραφή και ολοκλήρωση τη σύμβαση. δεν κατάφεραν όλα τα κράτη-μέλη που είναι ε, αρμόδια για θέματα που καλύπτει η Σύμβαση του Μαυρίκιου να συμφωνήσουν να εφαρμοστεί αυτή η σύμβαση στην αλλά η Προεδρία είναι δεσμευμένη για να υπάρξει πρόοδο στο σημαντικό αυτό φάκελο. Είναι μία από τι προτεραιότητέ μα και θέλουμε να προχωρήσουν οι συζητήσει του επόμενου 6 μήνε. Ε, διμερείς επαφές με αντιπροσωπείε ε, θα τι προωθήσουμε και θα τι συνεχίσουμε για να εξαλείψουμε τι ε, υπολείπουσες διαφορές και ενθαρρύνουμε όλα τα κράτη-μέλη να έχουν μια επικοδομητική στάση στο θέμα αυτό, ούτω ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να υπογράψει την σύμβαση για την σύμβαση του ενεργειακού κεφαλαίου. Έχουμε προχωρήσει με τη διατύπωση και με αναδιατύπωση της ε, επενδυτικής πολιτικής που είναι επιμερισμένης ευθύνη. Ε, η Ένωση και τα κράτη-μέλη ε, έχουν πραγματογνωμοσύνη στην προστασία των επενδυτών και γι' αυτό το Νοέμβριο του 2015 το Συμβούλιο καλωσόρισε την καινοτόμα προσέγγιση για να εξυγχρονίσει την προστασία των επενδυτών. Το Συμβούλιο σημείωσε την πρόθεση της Κομισιόν να εξετάσει αυτή την προσέγγιση και σε άλλες εμπορικές συμφωνίες όπου δει και να εργαστεί προς την δημιουργία ενός πολυμερούς ε, επενδυτικού δικαστηρίου ως τελικό στόχο. Επίσης, την δέσμευση να σεβαστούμε το, δικαίωμα μιας χώρας να ρυθμίζει σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της, της Σύμβασης Διαφάνειας σε διμερείς ε, συνθήκες. Η Προεδρία είναι απόλυτα δεσμευμένη στο στόχο της αυξημένης διαφάνειας ό,τι αφορά το σύστημα ε, διαιτητικής επίλυσης διαφορών επενδυτών κρατών. Δεν μπορούμε ως Προεδρία να ανακατευτούμε στι αρμοδιότητε των κρατών μελών εύκολα. Δεν μπορούμε να ξαναγκάσουμε τα κρατη να εφαρμόσουν τους κανόνες διαφάνειας της Φουνσιτράλ στις δικές τους διμερείς ε, συμφωνίες που έχουν συναυθεί πριν από την 1η Απριλίου του 2014. Ε, με αυτό το πλαίσιο όμω, με δεδομένο αυτό το πλαίσιο, εγώ ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε λύσει στο Συμβούλιο για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα ε, και από πλευράς Προεδρίας ε, εργαζόμαστε πάρα πολύ έντονα, ούτως ώστε να το, κάνουμε αυτό, να το καταστήσουμε αυτό πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σιτσού είναι ο επόμενος ομιλητής. Τσιτσού. η ομάδα του ΕΛΚΑ θεωρεί ότι η συμπερίληψη κανόνων για τη διαφάνεια στο πλαίσιο διεθνών συμβάσεων πέραν του ότι βελτιώνουν τη διαφάνεια στις ε, διαφορές έχουν και ως συνέπεια να δώσουν μεγαλύτερη αξιοπιστία στις συμφωνία. συνολικά. Διότι αυτά τα δύο στοιχεία για μας του ΕΛΚ είναι εξαιρετικά κεντρικά και σημαντικά. Απευθύνουμε λοιπόν προς το Συμβούλιο σήμερα ζητώντας ε, απαντήσεις που δόθηκαν ε, και που μόνο εν μέρη μας ικανοποιούν για αυτή την κατάσταση της επιβράδυσης που προκύπτει, διότι η Ένωση πρέπει να πρόκειται για την πρώτη σύμβαση, μεταρρύθμιση σύμβαση για τη βελτίωση των, ε, του, της επίλυσης των διαφορών. Όπως ξέρουν οι συνάδελφοι στην Επιτροπή, ότι η εναρμόνιση των κανόνων αυτών είναι βασικός κανόνας και προτεραιότητα για το μέλλον της αξιοπιστίας των εμπορικών διεθνών συμφωνιών όπου η Ένωση επενδύει και όπου η Ένωση αποτελεί ένα εγχείρημα που γίνεται με βασικές θεμελιώδεις ψηφίδες. Αυτή η ε, στασιμότητα μπορεί να ε, οδηγήσει σε αρνητικές επιπτώσεις. Η συμφωνία που γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή στηρίζεται στο, στον, στην ιδίως η Συμφωνία για την Ενέργεια στηρίζεται στην ε, σταθερότητα των ε, συμφωνιών. Οι κανόνες διαφάνειας ε, στους, στο πλαίσιο των, της διαιτητικής επίλυσης διαφορών μόνο μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο μπορεί να λυθούν. Ο κύριος Μάρτιν, πρόεδρε ευχαριστώ και ευχαριστώ την Προεδρία πρώτον που έμεινε εδώ και παρακολουθεί την συνεδρίαση για τις θετικές απαντήσεις και για το ναι, ναι, ναι. Ξέρουμε βέβαια τι σημαίνει ότι εσείς πρέπει να κάνετε και να κάνετε και να κάνετε στο επόμενο πλαίσιο, στο επόμενο διάστημα. Γνωρίζει το τι πρέπει να κάνει το Συμβούλιο στο ISDS. Εμείς δεν θέλουμε να συνεχίσει η Κομισιόν να χρησιμοποιεί μυστικές διαπραγματεύσεις. Εμείς ζητούμε μακροπρόθεσμα μια πιο πολυμερή λύση της επίλυσης διαφορών, αλλά ταυτόχρονα ζητούμε μεγαλύτερη διαφάνεια στις υφιστάμενες διατάξεις επίλυσης ε, διαφορών. Υποστηρίζουμε τις ε, προτάσεις ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα εφαρμόζονται στα υφιστάμενα ε, στι φυστάμενη συμφωνίε των κρατομελών και στο χάρτη ενέργεια. Ε, η δουλειά στο Συμβούλιο, το έργο στο Συμβούλιο δεν μπορεί να προχωρήσει, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Εμεί συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την ανάγκη να διευκρινιστεί ότι οι επενδύσει είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα και είναι κρίμα που οκτώ κράτη-μέλη υπέγραψαν μονομερό τη σύμβαση χωρί να περιμένουν την άδεια της Ένωσης. Αυτό δείχνει προς τα έξω ότι είμαστε ε, διαιρεμένοι, ανοργάνωτοι, ενώ χρειάζεται να έχουμε μια ισχυρή φωνή στο πλαίσιο αυτό. Επίσης ανησυχεί το γεγονός ότι ακούμε πως μέσα στο Συμβούλιο ε, κάποια κρατημέρια δεν υποστηρίζουν τους κανόνες διαφάνειας. Οι νέοι αυτοί οι κανόνες είναι ελάχιστες, ελάχιστα πρότυπα, ελάχιστες απαιτήσει για την Ένωση και θα έπρεπε να υποστηριχθούν ομόφωνα από το Συμβούλιο. Ζητούμε από το Συμβούλιο να εξοδίσει την Ένωση να υπογράψει τη σύμβαση του στο Μότο του Συνεφανωστή και στο Χάρτη ενέργεια και ζητούμε από τα κράτη-μέλη να, να, να επιτρέψουν την εφαρμογή των ίδιων κανόνων σε όλες τις μερικές συμφωνίες. Η Ένωση είναι ένας ε, ε, ε, ένας από τους φορείς που παίζει πρωταρχικό ρόλο στις επενδύσεις θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι η επένδυση είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης και να προχωρήσει στην, ε, στις συναφής επιπτώσεις. Η κυρία Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον αρμόδιο Υπουργό, ο παρέμεινε εδώ για να ακούσει τη συζήτηση. Αυτό είναι ένα απλό θέμα Μιλάμε πάρα πολλές φορές για τη διαφάνεια σε αυτό το κοινοβούλιο και πιστεύουμε στην αρχή της διαφάνειας. Μερικές φορές όμως είναι δύσκολο να αποδεχτούμε αυτά τα οποία μας λέει το Συμβούλιο και αυτή είναι μία από τις συγκεκριμένε τέτοιε περιπτώσεις. Είναι δύσκολο να δεχτούμε ότι το Συμβούλιο δεν έχει καταφέρει ακόμα να ξεπεράσει το διέξοδο το οποίο έχει δημιουργηθεί. Θα ήθελα να προσπαθήσω να καταλάβω γιατί εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η κατάσταση. Θα σα ρωτούσα αν έχετε αναλάβει ένα ενεργό ρόλο σε, στην επίλυση αυτού του αδιεξόδου. Μας είπατε ναι. Πολύ καλό τότε να σας ρωτήσω περισσότερες λεπτομέρειες. Τι ακριβώς κάνετε. Και ίσως μπορείτε να είστε λίγο πιο διάφανος σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις που λαμβάνουν χώρα μέσα στο Συμβούλιο σε σχέση με το πώς θα επιλύσετε το πρόβλημα αυτό. Είναι προφανές ότι όλα αυτά επηρεάζουν την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εξωκόσμο. Είναι λυπηρό το ότι 8 κράτη-μέλη αναγκάστηκαν να, κάνουν μονομερός, να προχωρήσουν μονομερός στο να υπογράψουν. Δεν φταίνε αυτοί, απλώς ήταν κάπως αδίμονα αυτά τα κράτη-μέλη. Λοιπόν, παρακαλώ το Συμβούλιο λοιπόν να κάνει τα απαραίτητα για να μπορέσει να υπάρξει μια λογική συμφωνία σε αυτό το τόσο λογικό μέτρο. Η κυρία Σουάκη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Κούντερ, χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια στη λήψη απόφασης και παροχή πληροφοριών σε σχέση με αυτά τα που αποφασίζουν. Αποφασίζει το Συμβούλιο. <clears throat> Αυτά ζητούμε και από την Επίτροπο Μάλστρομ στα θέματα του ISDS να γίνουν δημόσια τα σχετικά έγγραφα. Θέλουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και σε σχέση με τη Συμφωνία για τη Διαμεσολάβηση μεταξύ επενδυτών και κρατών η σύμβαση του ΟΗΕ εδώ έχει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη ε, διαφάνεια στους μηχανισμούς ISDS που όπως ξέρετε είναι πολύ αμφιλεγόμενοι. Είναι παράλογο λοιπόν για μένα το γεγονός ότι το Συμβούλιο που είναι αρμόδιο για περίπου 1.400 τέτοιους μηχανισμούς σε συμβάσεις Ευρω... συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κάνει τίποτα. Είναι απαραίτητο το Συμβούλιο να κάνει πραγματικότητα αυτή τη διαφάνεια. Η ίδια η Ολλανδία δεν έχει υπογράψει αυτή τη σύμβαση για μεγαλύτερη διαφάνεια παρά τις εκκλήσεις πολλών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Κάποιες χώρες όμως η Σουηδία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ιταλία έχουν υπογράψει τη συμφωνία αυτή. Τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς είναι πιο Έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς το πρόβλημα οφείλεται στο ίδιο το Συμβούλιο. Υπάρχουν πολλοί υπουργοί οι οποίοι εμποδίζουν τις προσπάθειες της Κομισιόν να επιτευχθεί μεγαλύτερη διαφάνεια. Δεν μπορείτε να υποχρεώσετε τα κάτι μέλη, μπορείτε να δώσετε όμως το καλό παράδειγμα ως Ολλανδική Προεδρία. Παρακαλώ, δείξτε πώς μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό δίνοντας το καλό παράδειγμα και πείθοντα κάποιε άλλε χώρε στο Συμβούλιο και ίσω μπορείτε να μα εξηγήσετε ποιε είναι οι χώρε οι οποίε εμποδίζουν την πρόοδο στο θέμα αυτό και τι θα κάνετε για να εξασφαλίσετε ότι θα επιτευχθεί μεγαλύτερη διαφάνεια για τα θέματα αυτά προς το όφελος όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Κύριο Σόλτς έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι, η υποσχόληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σύμβαση του ΟΗΕ θα βοηθήσει πάρα πολύ να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί σε σχέση με την χάρτα ε, και να μπορέσει επιτέλους να αναλάβει πραγματικά τις ευθύνες της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό εγώ υποστηρίζω τα ερωτήματα που τέθηκαν προς το Συμβούλιο. Το μόνο πρόβλημα όμως είναι η ίδια η Σύμβαση για τα ενεργειακά θέματα. Το 2004 έχει ξεπεραστεί ακριβώς και το ρεκόρ σε τέτοιες διαδικασίες ISDS που δίνουν πλεονεκτήματα στους ε, ε, επενδυτές των κρατών μελών με αδιαφανείς διαδικασίας διαμεσολάβησης. Η Ιταλία απειλείται συνέχεια με τέτοιες διαδικασίες επειδή έχει αποφασίσει να έχει την δική της λύση για τα ενεργειακά θέματα. Ακόμα και η Γερμανία έχει μια αρνητική εμπειρία από τα θέματα αυτά και πρέπει το Συμβούλιο να τα λάβει όλα αυτά υπόψη της. Μπλε κάρτα για σας κύριε Σόλτς, αν μπορείτε να απαντήσετε. Ο κύριος Κάσπαρη. Κάσπαρη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σόλτς, είπατε ότι υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κάνει προσφυγές κατά της ε, Γερμανίας λόγω της ε, σύμβασης αυτής. Η κολονία και το μόναχο όμω χρησιμοποιούν και αυτή αυτήν την ε, σύμβαση. Είναι αδιφάγες και αυτές οι εταιρείε που θα προσπαθούν να βγάλουν κέρδος από αυτή τη σύμβαση. Κύριο Σόλτς χωρίς μικρόφωνο. Δεν θεωρώ ότι εκεί το πρόβλημα. Εσείς και εσείς ακολουθείτε την λογική της, ε, του ISDS που μπορεί να οδηγήσει σε προσφυγές κατά των αρχών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Κάθε μέρα λοιπόν εφαρμόζεται αυτή η πρακτική η οποία χρησιμοποιείται προς ε, η απόκτηση μεγαλύτερου κέρδους. Φίντσου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το εμπόριο θα πρέπει να φέρνει οικονομικά ωφέλη και δεν θα πρέπει να είναι πολιτική. Και όμω εμεί χρησιμοποιούμε το εμπόριο για να προωθήσουμε την πολιτική μα ατζέντα. Αυτό κάνουμε και με τη Σύμβαση του Μαυρίκιου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει όλα τα κράτη-μέλη να υπογράψουν, ούτω ώστε η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να υπογράψει ε, για να εξυπηρετήσει τα δικά τη συμφέροντα, να καταστήσει το ISDS, τον πυλώνα τη εμπορική πολιτική. Η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση θεωρεί ότι το ISDS είναι θεμητό σύστημα, αλλά δεν είναι. Ε, ακυρώνει το εθνικό δίκαιο, έχει απορριφθεί από δύο επιτροπές του Κοινοβουλίου και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων του TTIP. Επίσης το, το μάχονται διάφοροι ευρωβουλευτές και παρόλα αυτά η Κομισιόν το θέλει ε, στις εμπορικές της διαπραγματεύσεις ε, και το έχει βάλει στο σχέδιο συμφωνίας με τον Καναδά. Ακούσαμε ε, τις ε, θριαμβολογίες, ε, διαφάνεια, προστασία των επενδυτών, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ενός αθέμητου και περί του συστήματος. Η Επίτροπος Μάστρομ είπε ότι τα κράτη θα πρέπει να υποστηρίξουν του ευρύτερου στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο βρισκόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ακυρώσουν, να απεμπολίσουν την ε, κυριαρχία του προ το συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μια μπλε κάρτα. Υπάρχει μια μπλε κάρτα. Από τον κύριο Μάρτιν. Είσαστε έτοιμος να απαντήσετε. Μπορείτε να μου πείτε πόσες ε, διμερείς ε, επενδυτικές συμφωνίες ε, ξέρετε παγκόσμια, τις οποίες έχουμε προσυπογράψει και εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο και που παραμένουν μυστικές. Γιατί αυτό δεν αφορά τις μελλοντικέ επενδυτικές συμφωνίες, τις παλιές, όπου πολύ σωστά είπε ο πρόεδρος, δεν γνωρίζουμε τι έχουν κάνει και κοστίζουν εκατομμύρια στερλίνες το φορολογούμενο κάθε χρόνο. Απάντηση. εκτό μικροφώνου. Όχι. Είναι η απάντηση. Όμως ισχύει ότι το ISTS το βάζουμε από την πίσω πόρτα, είναι απαράδεκτο. Οποιοδήποτε πιστεύει ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα των απλών ανθρώπων θα πρέπει να το ξέρει και θα πρέπει να δεχθεί το γεγονός αυτό. Κύριος Μπάλτσερ. Ευχαριστώ πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Πρόεδρε, όσοι έθεσαν την ερώτηση αυτή θέλουν να ε, πετύχουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπογράψει τη συνθήκη που επιτρέπει στους επενδυτές να στραφούν στην επίλυση διαφορών διαιτητικά. Η απόφαση αυτή είναι οριστική και η Ένωση δεν μπορεί να υπογράψει τη συνθήκη αυτή αν ε, παρεμποδιστεί από έναν συγκεκριμένο ρυθμό κρατών μελών. Όσοι που αμφισβητούν κάτι τέτοιο θέλουν να ζητήσουν από, το, την Προεδρία να ασκήσουν πίεση στα κράτη-μέλη αυτά. Η διαδικασία αυτή είναι κάπως ε, άδικη. Ακούσαμε κάποιους να λένε ότι η διαδικασία διαιτητικής επίλυσης διαφορών είναι παράνομη και επηρεάζει την, ε, και παρεμβαίνει στην εθνική κυριαρχία. Γιατί να υποστήριξουμε μια τέτοια διαδικασία όταν δεν έχει διαφάνει Ο κ. Κάσπαρη, επόμενο ομιλητή. Κυρία Πρόεδρε, η προστασία από τις απαλωτριώσει χωρίς αποχρόντα λόγο είναι ένα βασικό στοιχείο της ε, ε δημοκρατίας και δεν πρέπει κάποιος να βρίσκεται σε μειονεκτική θέση λόγω εθνικότητάς του τα επενδύει σε μια άλλη χώρα. Δυστυχώς, ένας από τους προηγούμενους ομιλητές από το Μεγάλη Βρετανία έφυγε από την και ήθελα να του πω ότι έχει υπογράψει η χώρα του πάρα πολλέ τέτοιε συμφωνίε. Η συνθήκη τη Λισαβόνα δίνει το δικαίωμα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα προστασία των επενδύσεων, <clears throat> αλλά να τροποποιήσουμε το σύστημα και δεύτερον θέλουμε να έχουμε διαφάνεια στα πλαίσια τη σύμβαση του ΟΗΕ. Γι' αυτό θα ήθελα να ξέρω από το Συμβούλιο να μου πει ποιε χώρε εμποδίζουν αυτήν την Γενική Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιοι είναι οι υπουργοί οι οποίοι αντιδρούν, σε ποια κόμματα ανήκουν και γιατί δέχονται, γιατί συνεχίσουν να εμποδίσουν την κατάσταση αυτή και δεν υποστηρίσουν την μεγαλύτερη διαφάνεια. Τι κάνει τελικά το Συμβούλιο, πότε θα εφαρμόσουμε οριστικά τα κράτη-μέλη τη ε, συνθήκη τη Λισαβόνα στον εμπορικό τομέα και θα αποδεχτούν ότι υπάρχουν πραγματικέ αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πώ μπορείτε να δικαιολογήσετε αυτή την αδράνεια του Συμβουλίου ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είπατε ναι, ναι, ναι στα τρία ερωτήματα. Εγώ βλέπω να λέτε τρει φορέ όχι. Πώ γίνεται κάτι τέτοιο. Επιτέλου κάντε αυτό το οποίο πρέπει να κάνετε και εξασφαλίστε ότι το, Ευρωπαϊκό, το Συμβούλιο θα αναλάβει πραγματικά τι ευθύνε του. Σίλβο Περέιρα. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη διαφάνεια στι διαιτητικέ διαδικασίε μεταξύ επενδυτών και κρατών μελών υπάρχει για δύο λόγου. Γιατί υπήρξε ένα σοβαρό πρόβλημα σε σχέση με τη διαφάνεια των συστημάτων διαμεσολάβηση και διαιτησία και διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε την ηγεσία στον αγώνα για μια σύμβαση η οποία θα έλυνε το πρόβλημα αυτό. Είναι ακατανόητο που τώρα που υπάρχει αυτή η σύμβαση και 8 κρατη την έχουν κυρώσει, εξακολουθούν να υπάρχουν ατέρμονες διαμάχες μέσα στο Συμβούλιο για να μην υπάρξει υπογραφή από την Ευρωπαϊκή Ένωση μια σύμβαση που ζήτησε η ίδια η Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Είναι απαράδεκτα λοιπόν αυτό και η καθυστέρηση στην εφαρμογή αυτής της σύμβασης θα έχει συνέπειε. Θέλω λοιπόν να παρακινήσω την Ολλανδική Προεδρία να τηρήσει τι δεσμεύσει που έχει αναλάβει η ίδια και να κάνει τι πρωτοβουλίε που απαιτούνται, όχι μόνο για να πει τα κράτη-μέλη να υπογραμμίσουν, να υπογράψουν αυτή τη σύμβαση, αλλά για να εξασφαλίσει ότι αυτοί οι νέοι κανόνε θα εφαρμόζονται στην χάρτα ενέργεια που περιλαμβάνει ένα σύστημα ε, επίλυση διαφορών με μεγαλύτερη διαφάνεια. Κυρία Σάντσερ καλή Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι προφανές πως υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα στα ISDS. E Η έλλειψη διαφάνειας είναι το μεγαλύτερο, αλλά όχι το μόνο. Το γεγονός ότι πολλά κράτη δεν δέχονται ούτε καν αυτό πρέπει να μας κάνει να καταλάβουμε ότι κάτι έγινε πολύ άσχημα. Είναι καιρός να αλλάξουμε την κατάσταση. Ξεκινάμε με τη διαφάνεια, αλλά πρέπει να πάμε παραπέρα. Κάθε κομμάτι του μηχανισμού αυτού είναι ε, επίφορο σε κατάχρηση από πλευρά ε, ε, επενδυτών. Το γεγονό ότι υπάρχει ρήτρα μη διάκριση ή ότι οι δικαστέ είναι και ταυτόχρονα και δικηγόροι. Χρησιμοποιώ τα λόγια του Άλφρεντ Τεσάγια, ειδικού ε, εισηγητή του ΟΗΕ, που αναφέρει ότι τα τελευταία 25 χρόνια οι διημερεί συμφωνίε με ISDS υπονόμευσαν τι βασικέ αρχέ των Ηνωμένων Εθνών, την κρατική κυριαρχία, τη δημοκρατία και το κράτο δικαίου. Ο, ο, ο παρατηρητή αποκτά μια ε, ηθική, ε, έναν ηθικό ύλικο. Η ύπαρξη των ISDS επιτίθενται ευθέω στα, στα θεμέλια τη δημοκρατία. Κυρία Μπεγγίν, ευχαριστώ Πρόεδρε. Μέχρι τώρα, 127 περιπτώσεις ISDS ε, ε, έχουν ε, μονογραφηθεί από πολλές πολυεθνικές και έχουν επιφέρει 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ και ακολουθούν άλλα 30 δισεκατομμύρια. Δεν έχουμε ιδέα πόσες πώς έχουν δοθεί μετά από φιλικές ε, συναλλαγές ε, στη Γερμανία, στην Πολωνία. Πέρα από αυτά τα νούμερα δεν λαμβάνουμε υπόψη πολλές άλλες μυστικές υποθέσεις. Για να αποφύγουμε αυτή την κατάσταση υπάρχει μια σύμβαση του ΟΗΕ που υποχρεώνει τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών που αφορούν τις περιπτώσεις ISDS που είναι εξελίξει. Μια σύμβαση ε, που όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλά κράτη δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη. Αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα, ειδικά στην ενεργειακή χάρτα, και που δημιουργεί ε, και που σχετικά υπάρχουν πάρα πολλές ε, διενέξεις. Ε, εμείς είμαστε κατά ως Cinque Stelle, γιατί θέλουμε κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες, τη διαφάνεια. Ο κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Κομισιόν, το Συμβούλιο, καθώς και τα κράτη-μέλη και οι διεθνείς οργανισμοί θα πρέπει να ανησυχούν και να προσπαθούν να παγιώσουν ένα οικονομικό πλαίσιο που θα εξασφαλίσει ασφάλεια των επενδύσεων και του διεθνούς εμπορίου. Να υπάρχει ένα εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο για ε, δίκαιη επίλυση των διεθνών διαφορών. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα αυξήσουμε την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Σε αυτό το πλαίσιο εκτιμούμε τις προσπάθειες που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κομισιόν για το δίκαιο του διεθνούς εμπορίου που προσπαθεί να εισαγάγει την έννοια της διαφάνειας όλη αυτή τη διαδικασία. Υιοθετώντα την ε, σύμβαση του ΟΗΕ για την ε, διαφάνεια σε, στη διαιτητική επίλυση διαφορών επενδυτών κρατών βάσει συνθήκης. Αυτή η σύμβαση θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ασφάλεια των επενδύσεων, οικονομική ανάπτυξη στα κράτη-μέλη και ουσιαστική αύξηση των θέσεων απασχόλησης. Παράλληλα, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα μεμονωμένα να υπογράψουν μια σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ε, διμερείς επενδυτικές συμφωνίες που έχουν υπογράψει στο παρελθόν. Δυστυχώς, οι διαπραγματεύσεις ε, για το τι που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα δεν, δεν εξασφαλίζει ε, τις απαιτούμενες θετικές εξελίξεις λόγω ακριβώς της διάταξης SDS. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε κάποιους διαδικαστικούς κανόνες σε διεθνές επίπεδο για να εξασφαλίσουμε αυτή τη διαφάνεια ε, από την αρχή ως το τέλος της διαδικασίας διατησία. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε και ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο και ευχαριστώ τον Υπουργό. Σε πολλές περιπτώσεις είχα αντιταχθεί στα ιδιωτικά δικαστήρια επίλυση διαφορών, αλλά το ISDS υπάρχει χάρη σε χιλιάδες συμφωνίες επενδύσεων. Οι επενδυτές της δικής μου χώρας χρησιμοποιούν συχνά τους μηχανισμούς αυτούς αυτό είναι, αυτός είναι ο λόγος τον οποίο είμαι υπέρ μιας μεγαλύτερης διαφάνειας στις συμβάσεις αυτές ακριβώς επειδή δουλεύουμε για μια καλή εναλλακτική στο ISDS. Πρέπει τις αποφάσεις αυτές να τις ε, βγάλουμε από τις κλειστές πόρτες, να μπει το φως της μέρας να υπάρξει μια κινητικότητα στο φάκελο αυτό και από πλευρά Συμβουλίου. Μιλάμε τώρα για το χάρτη ενέργεια, αλλά το θέμα είναι ευρύτερο. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να ξέρουμε πώς θα μπορέσουμε να έχουμε ανοιχτή και διάφανη προστασία των επενδύσεων. Η κυρία Μόσκα και μετά το Κατσιδιάη εκφραστήκαμε σαφώς το θέμα της διαφάνειας. Είναι βασικός πυλώνας του τρόπου με τον οποίο καταλαβαίνουμε το πώς γίνεται η εμπορική πολιτική της κοινότητας και είναι ο μόνος τρόπος για να έχουμε καρποφόρες επαφές και συνεργασία με τους εταίρους και με την κοινή γνώμη. Γι' αυτό θεωρώ κρίμα το ότι χρησιμοποιήθηκαν διαδικαστικές, ε, ε, διαδικαστικά επιχειρήματα για την ε, καθυστέρηση της επίλυσης διαφορών και διότι πολλές, ε, πολλά κρατημέλη δεν έχουν επικυρώσει τη σύμβαση. Αντιλαμβάνομαι τα όρια του Συμβουλίου. Ωστόσο, εμείς, ε, αντίθετα από άλλους συναδέλφους, θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει παρέμβαση όλων των θεσμικών δρόντων για να διευκολυνθεί η επίλυση του προβλήματος. Είναι μια στιγμή κλειδί για την επίλυση της διαδικασίας διαιτητικής επίλυσης διαφορών. Αυτό δείχνει και αν θα είμαστε ή όχι σαν Συμβούλιο κυρίως όριμοι για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Διαδικασία Catch the Eye. Δύο άτομα έχουν ζητήσει το έργο. Κύριος Μαριάς πρώτα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συζητούμε για την ε, διαιτητική επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών, τη γνωστή ISDS καθώς επίσης και για τα ζητήματα διαφάνειας που προκύπτουν κατά τη λειτουργία της. αρχικά αυτό που επιτυγχάνει μέχρι στιγμής το σύστημα isds είναι να επιτρέπει στις πολυεθνικές επιχειρήσεις να προσφεύγουν εναντίον συγκεκριμένων κρατών για ζημιές τις οποίες υπέστησαν οι επιχειρήσεις αυτές κατόπιν αποφάσεως δημοσίας πολιτικής. καταργείται δηλαδή το υπάρχον σύστημα δικαστικής προστασίας και οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα μέσω των isds να αποζημιώνονται αδρά από τα κράτη παράλληλα προκειμένου να υπάρξει διαφάνεια για τις isds η ευρωπαϊκή ένωση οφείλει να ενσωματώσει τα πρότυπα διαφάνειας της επιτροπής ηνωμένων εθνών για το διεθνές εμπορικό δίκαιο σε όλες τις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες συμπεριλαμβανομένων και των συνομιλιών με τις ηνωμένες πολιτείες σχετικά με την ttip ανάμεσα στις δράσεις που προτείνει η επιτροπή των ηνωμένων εθνών για την επίτευξη της διαφάνειας περιλαμβάνεται και η δημοσιοποίηση των διαπραγματευτικών κειμένων της ευρωπαϊκής ένωσης καθώς επίσης να είναι ανοιχτές προς το κοινό οι σχετικές ακροάσεις. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα εξ αρχής να εκφράσω την θετική μου άποψη για την πρόθεση αυτή να υπάρξει υπογραφή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών και να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια. Ελπίζω και περιμένω από την Ολλανδική Προεδρία να πείσει τα κατημέλη να υπογράψουν αυτήν την ε, σύμβαση μέσω της οποίας θα μπορέσει να γίνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση προς υπογράφων μέλος. Γιατί ο μηχανισμός ISDS περιλαμβάνει πολλά προβλήματα και είναι απαραίτητο να γίνει μια προσπάθεια επίτευξης μεγαλύτερης διαφάνειας <clears throat> στις εμπορικές σχέσεις. Η χώρα μου έχει υπογράψει μια ε, συμφωνία, τη συμφωνία αυτή για τα ενεργειακά θέματα και εγώ είμαι πεπισμένος ότι σε αυτό το σημείο μπορεί να θυγούμε διότι πήραμε μια τέτοια θέση πρέπει να έχουμε το μεγαλύτερο επίπεδο ε, για το καλό μας. Κύριε Κούντερας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ακούω με πολύ ενδιαφέρον τις απόψεις σας για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμα αυτά που είπατε για να μπορέσουμε να ξέρουμε μια επαρκή λύση και μια λύση που θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προσχωρήσει στη σύμβαση για την ε, διαφάνεια στην, ε, στις διαμεσολαβήσεις αυτού του είδους. Όταν είπα στην αρχή ναι, ναι, ναι, βλέπω ότι το συμπέρασμα από εσά ήταν να κάνουμε, να κάνουμε και να κάνουμε. Αυτό είναι λογικό να περιμένετε ότι θα πρέπει να υπάρξει δράση από εμάς αλλά από τις περισσότερες απόψεις που άκουσα είναι φανερό ότι δεν υπάρχει διαφωνία γιατί η διαφάνεια είναι πάρα πολύ σημαντική για την Προεδρία μας. Θέλουμε να έχουμε πιο απλή και πιο αξιόπιστη νομοθεσία. Ανέφερα και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου πέρσι. Η Προεδρία μας είναι προσφυλωμένη στην επίτευξη πρόοδου για αυτό το σημαντικό θέμα. Είναι από τα θέματα προτεραιότητας για τα οποία θέλουμε να προχωρήσουμε το επόμενο εξάμεινο και ζητάμε να υπάρξουν επιμέρειες επαφές με τις εμπλεκόμενες εθνικές αντιπροσωπείε, Θα συνεχιστούν αυτές για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις διαφωνίες που υπάρχουν. Δεν έχουμε ακόμα υπογράψει λοιπόν τη σύμβαση του Μαυρικίου. Είμαστε 100% υπέρ της διαφάνειας που περιλαμβάνεται στη σύμβαση αυτή βέβαια, αλλά υπάρχουν διαφορές απόψεων όπως αναφέρθηκε και από εσά <clears throat> από την σοσιαλιστική ομάδα. Κάποιοι θεωρούν ότι δεν πρέπει ένα κράτο μέλο να ζητά έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να προσυπογράψει αυτή τη σύμβαση. Εμεί αποφασίσαμε να περιμένουμε, αλλά και εμεί αρχίσουμε να νιώθουμε ανυπομονησία, γιατί θέλουμε αυτή η διαφάνεια να εξασφαλιστεί και γι' αυτό είναι λυπηρή η κατάσταση που επικρατεί στο Συμβουλίο. Αυτό θα συμφωνήσω και με τον κύριο Λάγκε, δίνει μια αρνητική εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης περιμένουμε το αποτέλεσμα της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τον μεικτό χαρακτήρα ορισμένων συμφωνιών. Πρέπει να λάβουμε λοιπόν την άποψη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την κατανομή ε, αρμοδιοτήτων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και 100 μελών για τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου με την Σιγκαπούρη και ελπίζουμε ότι θα γίνει και αυτό πραγματικότητα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν το συνολικό είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουμε να βρούμε κάποια λύση στο Συμβούλιο για αυτό το σημαντικό θέμα και σίγουρα εργαζόμαστε για να το κάνουμε αυτό πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Πέρα τη συζήτηση.